την έκθεση της κυρίας Ένης Πλάσερ για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης, ανείχνευσης και, ε, και καταπολέμησης τρομοκρατίας. Γνωρίζετε ότι από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολλοί άριθμα μέτρα έχουν ληφθεί σχετικά με αυτό το θέμα. Η απαρτίζεται από άμεσα ερετούς εκπροσώπους των πολιτών. Είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για τα δικαιώματα των πολιτών λοιπόν και πρέπει ως θεματοφύλακες αυτών των δικαιωμάτων να διαδραματίσουμε το ρόλο μας. Είναι απόλυτα σαφές αυτό και πρόκειται για την πρωτογενή μας πρωταρχική αρμοδιότητα. Γνωρίζουμε όλοι λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι το θέμα του SWIFT για τελείως διαφορετικούς λόγους βέβαια και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια ισορροπημένη αντιμετώπιση των ε, σχετικών θεμάτων μια εξισορρόπησή τους. Ε, η συνθήκη της Λισαβόνας άρχισε να ισχύει. Ε, ήδη τον Νοέμβριο 2009 εστράφη προς τον κύριο Πρωθυπουργό Ράινφελτ και απίφθηνα μια επιστολή στον τότε προεδρεύοντα υπό τη Σουηδική Προεδρία με την παράκληση να αναβληθεί η λήψη απόφασης και να αναμένει το Συμβούλιο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις συνθήκες της Λισαβόνα. Αυτό όμως δυστυχώς δεν έγινε. Στις 30 λοιπόν Νοεμβρίου το Συμβούλιο έλαβε την αντίστοιχη απόφαση επί του SWIFT και εγκρίθηκε το SWIFT. Στις 20, 21 Δεκεμβρίου επέστειλα μια νέα επιστολή εκ νέου προς τον κύριο Πρωθυπουργό Ράιντφελτ και έλεγα ότι αναμένει δύο πράγματα το Κοινοβούλιο. Αφενός να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότησή μας όσον αφορά την εντολή για την συμφωνία αυτή και δεύτερον πλήρως να ενημερώνεται η Ευρωβουλή σε σχέση με μελλοντικούς γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ. ΕΕ. Μια αντίστοιχη επιστολή απίθυνα επίσης και στον Πρωθυπουργό κύριο Θαπατέρο προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά αυτό το εξάμεινο. Και έτσι επανέλαβα αυτά τα αιτήματά μου και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Ταυτόχρονα απίθυνα μια παρόμοια επιστολή προς τον κύριο Μπαρόζο. Και ήμουνα και ήρθα σε επαφή με την κυρία Χίλαρη Κλίντον και άλλους εκπροσώπους ε, της ε, Αμερικανικής Διοίκησης των Αμερικανικών Αρχών και έλαβα και αντίστοιχη τοποθέτηση από πλευρά των ΗΠΑ. Είναι λοιπόν γνωστά σίγουρα αυτά και τα έγγραφα είναι σε όλους διαθέσιμα. Είναι γνωστά αυτά και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναδήποτε στιγμή μπορεί κανείς να εξοικειωθεί με αυτά τα θέματα αν χρειάζεται. Πρέπει να λάβουμε με υπεύθυνο τρόπο μια απόφαση και να μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι. Η σημερινή συζήτηση αυτό το σκοπό εξυπηρετεί. Γι' αυτό είναι μια τόσο σημαντική συζήτηση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που εκπρόσωποι του Συμβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παρόντες και συμμετέχουν, θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Θα ακολουθήσει λοιπόν η συζήτηση από πλευράς μας με τις παρεμβάσεις μας ως πιστή εικόνα του πώς αντιδράει η Ευρωβουλή και τοποθετείται. Τώρα, in media stress, περνάμε κατευθείαν στο θέμα, στην καρδιά του, στον πυρήνα του θέματος. Πρώτα, η κυρία εισηγήτρια Ζανίν Πλασέτ Φλένης ε, έχει τον λόγο, παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω λέγοντας ότι και εγώ είμαι υπέρ μιας ισχυρής ένωσης που να μπορεί να αντιμιλήσει αν χρειάζεται στη ΣΥΠΑ. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα του πώς θα πρέπει να συνεργαστεί στην καταπολέμηση της τραμακρατίας η Ένωση με τις ΗΠΑ. Χωρίς αμφιβολία η προβλεπόμενη ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητη, αλλά θα ήθελα να είναι σαφές ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να, έχουν, πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι και καταπολεμάται η ανασφάλεια και γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Το Συμβούλιο δυστυχώς δεν το είπε αυτά ρητός. Βλέπετε ότι η ισχύουσα, η προτινόμενη λοιπόν νομοθεσία δεν αποτελεί ενίσχυση της ε, προηγούμενης. Εμείς αντίθετα θέλουμε να εξεταστούν και από Ευρωπαίους τα στοιχεία που θα τεθούν σε Αμερικανούς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις λεγόμενες limited requests γιατί πρόκειται για παραβίαση των βασικών αρχών της νομοθεσίας της Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αναλογικότητα κλπ. Πάντοτε πρέπει να είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο δεν σκοπεύει απλώς παθητικά να λάβει γνώση των αποφασισμένων από το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε συνεχώς υποσχέσεις για το αύριο. Θέλουμε από τώρα δεσμεύσεις. Μέχρι τώρα δυστυχώς το Συμβούλιο ό,τι και να λέμε εμείς δεν έχει αντιδράσει. Δηλώνει ότι θα υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά δεν έχει πράξει τίποτα για να γίνει η προστασία αυτή απτή. Δηλώνει ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά γιατί κρύβεται πίσω από την Κομισιόν, αφού εκείνο θα εγκρίνει τελικά τις οδηγίες για τις διαπραγματεύσεις. Γιατί δεν έχει ακόμα συζητήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν συζητάει καθόλου το ότι με αυτόν τον τρόπο η Ένωση χορηγεί δικαιοδοσίε στη ΣΥΠΑ για τον έλεγχο των δεδομένων. Πρέπει τα δεδομένα που έχουν οι ΙΠΑ να τα έχουν και οι αρχές της Ένωσης ώστε κάποτε να καταλήξει σε αυτόνομη δική της δυνατότητα ελέγχου. με ανάλογο τρόπο με την οδηγία για την προστασία δεδομένων για τα τηλέφωνα. Επομένως το Συμβούλιο δεν παίζει το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει. Η μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων δεν είναι αναλογική και το Συμβούλιο δεν προβλέπει καμία ενωσιακή λύση για το πρόβλημα. Πέστε μου λοιπόν κύριε Προεδρεύοντα, πώς είναι δυνατόν να πω σε 500 εκατομμύρια πολίτες ότι τα δεδομένα τους δεν θα τύχουν σεβασμούς απλώς και μόνο γιατί το Συμβούλιο δεν έχει μία συνεπή στάση. Θα ακούσω ό,τι έχετε να μου πείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια. Και τώρα εξ ονόματος του Συμβουλίου θα λάβει τον λόγο ο Προεδρεύων κύριος Ρουμπακάβα παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή την παρέμβασή μου με μια αναμφίσιμη τοποθέτηση από πλευράς μου. Η Ισπανία υποστήριξε στεναρά και με κάθε τρόπο κάθετα την συνθήκη Λισαβόνα από την πρώτη στιγμή και το έκανε με την πεποίθηση ότι γνωρίζοντα ότι με την δρομολόγηση τη νέα συνθήκη θα συνεπαγόντουσαν πολλά νέα πράγματα στην προσέγγιση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσον αφορά τους ίδιους τους πολίτες μας. Είναι ένας στόχος που αναθέτει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την Ευρωβουλή συνθήκη, στο πρωταγωνιστικό του ρόλο, στη δράση του όσον αφορά τον χώρο πολιτικών ελευθεριών, τη δικαιοσύνη και εσωτερικών θεμάτων. Έτσι η συνθήκη θέλει να διευκολύνει την προσέγγιση μεταξύ θεσμικών οργάνων και πολιτών. Να ξεκινήσω λοιπόν αυτή μου την παρέμβασή μου διασφαλίζοντας ενώπιον ημών, κύριοι Ευρωβουλευτές, τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε από κοινού. Πιστά να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και με την Ευρωβουλή και να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο την Προεδρία μας. Είναι αυτό ένα συμπέρασμα από την Ισπανική Προεδρία που γεννάται από τη στεναρή δέσμευσή μας υπέρ της συνθήκης Λισαβόνας και των στόχων της. Το Συμβούλιο συμμερίζεται επίσης με αυτό το σώμα, την Ευρωβουλή, το μέλημα και την ανησυχία να διασφαλιστεί η ασφάλεια συνολικά των Ευρωπαίων πολιτών. Η ασφάλεια Ω ως εγγύηση για πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Αυτή είναι η αρχή που εμπνέει τον κοινό μας αγώνα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οποιασδήποτε μορφής τρομοκρατίας. Όπως έλεγε και το ψήφισμα της 17ης Σεπτεμβρίου του Σώματος και αναφέρω ως παράθεμα, το Σώμα, η Ευρωβουλή, με σθένο ακολούθησε τον στόχο καταπολέμηση τη Τρομοκρατία και έχει τη στεναρή πεποίθηση ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί μια ισορροπία, σωστή ισορροπία μεταξύ των μέτρων για την ασφάλεια και τη προστασία των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. τέλο παραθέματο. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με αυτό το παράθεμα, με αυτήν την τοποθέτηση. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα ήθελα να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Ένα νέο πλαίσιο. Το πλαίσιο τη συνθήκη ανοιχτής και ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και ένα μέλημα κοινό που δεν είναι πλέον καινούριο η καινοτόμο, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά υποσεβασμό των αρχών της αναλογικότητας και της ε, αποτελεσματικότητας, που είναι ταυτόχρονα η εγγύηση, τα ειχέγγυα για πλήρη δράση και αποτελεσματικότητα. Και έτσι απορρέει, Πρόεδρε, ότι η διεθνή τρομοκρατία έθεσε νέε προκλήσει ενώπιον των κοινωνιών μα. Πρόκειται και για νέα μορφή τρομοκρατία ε, που έχει ε, διάχυτη μορφή και παγκόσμια δρά. Έτσι λοιπόν η εκρίζωση αυτού του φαινομένου τίθεται σε παγκόσμια κλίμακα. Εδώ υπάρχουν δομές, ε, οι ελαστικές δομές μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο με μια ειδική προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης μας οδήγησαν αυτά τα πράγματα στο να μεγεθύνουμε και να μεγιστοποιήσουμε την εγρήγορσή μας. Πρόληψη λοιπόν, συντονισμός, πληροφόρηση, ενημέρωση. Είναι οι έννοιες, οι τρεις αυτές έννοιες άξονες της στρατηγικής μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια απειλή. Όλες οι χώρες προσπαθήσαμε λοιπόν να συντονιστούμε με τον καλύτερο τρόπο εσωτερικά και εξωτερικά για να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι και περισσότερο ενημερωμένοι για να συνεργαστούμε εν τέλει με εκείνους ε, που έχουν ακριβώς ενστερνιστεί τους ίδιους στόχους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και από πλευρά μας ε, έχουν πολλαπλασιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ομάδες ε, και οι ανταλλαγές στοιχείων και οι αναλύσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για τη διαβίβαση χρηματοοικονομικών δεδομένων, θέμα που εξετάζουμε σήμερα, η ανταλλαγή ε, δεδομένων χωρίς συμφωνία λειτουργούσε εδώ και χρόνια και μάλιστα χωρίς διακοπή. <clears throat> Όταν παρουσιάστηκα πριν από κάποιες εβδομάδες στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αρκετοί ευρωβουλευτέ με ρώτησαν για αυτή την ανταλλαγή στοιχείων. Ήταν μια απόλυτα σκόπιμη ερώτηση που στη δεύτερη έκθεση του, ε, από πλευρά δικαστού Γκουγιέρ είχε καλυφθεί και που διαβιβάστηκε στο σώμα και ως παράθεμα αναφέρω. Κατά τη διάρκεια του 2009 το TFTP ήταν ένα μέσο υψηλής αξίας για να ε, μείνουμε στην χαρτογράφηση της τρομοκρατίας. Να συμπληρώσουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία χρειαζόντουσαν για τις ανακρίσεις και τις ε, έρευνες, για να εντοπίσουμε την ταυτότητα των υπόπτων, για να γεωγραφικά τοποθετήσουμε και εντοπίσουμε, ώστε να μπορούμε να ανακαλύψουμε νέους υπόπτους και να αποφύγουμε νέες επιθέσεις τρομοκρατών. Τέρμα παραθέματος εδώ και προσθέτω όχι μόνο το 2009, αλλά επίσης και πιο πριν. Στη ΣΥΠΑ, στην Ευρώπη και παντού, παγκόσμια. Στη Βαρκελόνη τον Ιανουάριο του 2008, στη Γερμανία <clears throat> το 2007 στο Λονδίνο μετά από τις επιθέσεις της 7 η Ιουλίου στις έρευνες της 11ης Μαρτίου στις τρομοκρατικές απόπειρες στην Μαδρίτη, στις δολοφονίες της Συμπαγκόγκ ή τις τρομοκρατικές βομβιστικές απόπειρες στο Μαλί. Αυτά είναι παραδείγματα που αναφέρει ο δικαστής στην έκθεσή του. Η ανταλλαγή λοιπόν στοιχείων έδωσε θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή επέτρεψε να αποφύγουμε τέτοιες ε, απόπειρες, να αποφύγουμε να προλάβουμε τέτοιες επιθέσεις, να μπορέσουμε να, διώξουμε, να καταδιώξουμε τους ε, τρομοκράτες ε, μετά από απόπειρες ή και πριν από αυτές έχοντας προλάβει τις επιθέσεις. Σε σχέση με το SWIFT που όπως αναφέρθηκε το 2007 η ανάγκη της αλλαγής δεδομένων αληθεύει ότι αυτός ο στόχος δεν υλοποιήθηκε πριν, μέχρι πριν από λίγους μήνες. Έπρεπε να αναθεωρηθούν τα πρωτόκολλα σε σχέση με τη λειτουργία της ανταλλαγής των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Έπρεπε αυτό να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγκρίθηκε η εντολή το 2009 και έπρεπε να ακαλύψουμε την περίοδο αβεβαιότητα μέχρι την έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Είναι γνωστό αυτό το οποίο συνέβη στη συνέχεια. Υπεγράφει μια προσωρινή συμφωνία για εννέα, ε, εννέα περίοδο που πρέπει να επικυρωθεί από το Σώμα, από την Ευρωβουλή. Μια συμφωνία προσωρινή. Εννέα μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων η Ευρωβουλή θα έπρεπε να θεσπίσει μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευση. Αυτό το σώμα, η Ευρωβουλή, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον από κοινού, για να υπάρξει η διατύπωση μια τελική καθοριστική συνθήκη. Αυτή ήταν η απόφαση. Πιθανόν να μην ήταν η καλύτερη, αλλά πρέπει να καταστεί σαφέ ότι η συνθήκη ad referendum, η συνθήκη αυτή, η συμφωνία που συζητάμε σήμερα, είναι εκείνη που πρέπει και να καλύπτει την ε, ασφάλεια των ιδιωτικών προσωπικών δεδομένων καλύτερα από τα πρωτόκολλα μέχρι τότε. Και αυτό επειδή αυτή η προσωρινή συμφωνία έχει πρόσθετες εγγυήσεις και εχέγγυα. Μεταξύ άλλων, θέματα που είχαν υποβληθεί ως συστάσεις από την Ευρωβουλή και από, τον, ε, από πλευράς ε, ε, εισήγησης της Ευρωβουλής. Εδώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου πλήρως έλαβε υπόψη και κάλυψε τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωβουλή οι επιστολέ που απεστάλησαν από τον πρόεδρο τη Ευρωβουλή, καθώ επίση και η έκθεση που συντάχθηκε από την κυρία Χένι Φλάσερτ, που ψηφίστηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών την 4η Φεβρουαρίου. Γι' αυτόν τον λόγο ενέκρινε το Συμβούλιο και απέστειλε στο Σώμα εχθέ ένα σημείωμα του οποίου τα σημαντικότερα στοιχεία θα ήθελα να συνοψίσω. Πρώτον, δέσμευση του Συμβουλίου να εντάξει πλήρω μια τελική συνθήκη σε μια τελική συνθήκη τα ειχέγγυα τη ε, εγγυήσει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καλύτερε προποθέσει για την ανταλλαγή των στοιχείων με τι εθνικέ αρχέ και με τρίτε χώρε. Και είναι αυτονόητο επίση βέβαια τι εγγυήσει, να ενισχύσουμε τι εγγυήσει που εμπεριέχονται στην ενισχύ συνθήκη και που πρέπει να ενισχυθούν στην καθοριστική τελική συνθήκη με αυστηρό περιορισμό των στόχων τη χρήση αυτών των στοιχείων και απόλυτη απαγόρευση άντλησης ε, ε, στοιχείων, εξόριξης στοιχείων ε, για άλλους σκοπούς. Εν τέλει, το Συμβούλιο μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, μετά από τη νέα, την έναρξη ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, δεσμεύεται να εκπονήσει μια διοργανική συμφωνία για μια πιο ελαστική δυνατότητα προσέγγισης σε σχέση με αυτά τα δεδομένα όσο αφορά τα διεθνή πλαίσια. Εδώ θέλω στεναρά να πω ότι η Ισπανική Προεδρία δεσμεύεται απόλυτα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και του όρου τη και με τη θεμελιώδη χάρτα, των, ε, ε, με τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα με το άρθρο 8 και επομίζεται επίση και τα συμμερίζεται τα ε, νόμιμα μελήματα που έχουν εκφραστεί από την Ευρωβουλή. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι η δέσμευση που μόλις διατύπωσα είναι εφικτός και μπορεί να λειτουργήσει στην επιστολή όσον αφορά και την Υπουργό Εξωτερικών κυρία Χίλαρη Κλίντον και τον κύριο Υπουργό Οικονομικών Timothy Γκέιτερ δεσμεύονται να υπάρξει κάλυψη των εγγύσεων των εχεγγύων όπως το μέλημα το οποίο εξεφράστηκε από την Ευρωβουλή κατά το παρελθόν. Είναι λοιπόν δυνατόν κυρίε και κύριοι η διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας που εξετάζουμε και συζητούμε σήμερα στη διαδικασία αυτή έγκρισης το Συμβούλιο να μην έκανε τα πράγματα με τον καλύτερο, βέλτιστο τρόπο. Όμω, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι το ότι σε αυτή τη διαδικασία το Συμβούλιο έμαθε πολλά πράγματα. Και σε αυτή την ε, ε, πράξη τώρα σημειώνει απόλυτα και λαμβάνει υπόψη τι ανησυχίε και τα μελήματα τη Ευρωβουλής στο Συμβούλιο. Όπω σήμερα η συμφωνία που εξετάζουμε και συζητούμε και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η βελτίωση υπέρ τη ασφάλεια των πολιτών μα, παγκόσμια αλλά και στην Ευρώπη ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προεδρεύοντα. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω εδώ κάτι, κάτι που προηγούμενα προανέφερα. Εγώ μία γραπτή απάντηση έλαβα όσον αφορά τις επιστολές μου προς το Συμβούλιο και διένυμα προς τις κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες ε, του σώματος αυτές ε, τις επιστολές. Τοποθετείτε εκεί το Συμβούλιο στα, ε, στις προσδοκίες μας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά κύριε Προεδρέμοντα για αυτή την δήλωση, τις επεξηγήσεις που δώσατε και για αυτή την τοποθέτηση όσον αφορά το Συμβούλιο. Τώρα, εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα λάβει τώρα τον λόγο η κυρία Επίτροπος ε, Σεσίλια Μάλστρομ. Παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κύριε Προεδρεύοντα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, για εχθές που μας δώσατε και σε μένα μαζί την ψήφο πιστοσύνη σας και εγκαθιδρύσατε τη νέα επιτροπή. Είναι η πρώτη μου μέρα δουλειά λοιπόν, αλλά είμαι ευγνώμων που μπορώ σήμερα να συζητήσω μαζί σα το σημαντικό θέμα τη ε, αποστολή στοιχείων στη ΣΥΠΑ με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, και στην συνεργασία μας στο πρόγραμμα νύχνευσης χρηματοδότησης τρομοκρατίας, το TFTP. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση να συνδυάσουμε την ε, διαβίβαση στοιχείων με την προστασία αυτών. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής, και ένας από τους στόχους ήταν να διασφαλίσουμε την, ε, την ε, εφαρμογή με βάση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2009. Θέλουμε να ενισχύσουμε το τμήμα προστασίας των δεδομένων όταν θα διαπραγματευτούμε την μακροπρόθεσμη ε, συμφωνία, δηλαδή ιδιαίτερα τις ισχυρότερες εγγυήσεις σε σχέση με την νόμιμη επεξεργασία στοιχείων και τη διαγραφή των στοιχείων. Η έκθεση αυτή ήταν διαθέσιμη για τους βουλευτές την περασμένη εβδομάδα και αυτό δείχνει τη σημασία του TFTP και την αξία της έρευνας ε, κατά της τρομοκρατίας. Η έκθεση για το TFTP έχει εντοπίσει, ε, ε, μάλλον αναφέρει πως το TFTP έχει ήδη εντοπίσει ύποπτους τρομοκράτες στα κράτη-μέλη μας και τονίζει πως το TFTP είναι πολύτιμο και ότι οι αξιόπιστες πληροφορίες είναι απαραίτητες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ζητά συγκεκριμένα παραδείγματα και νομίζω το Συμβούλιο αναφέρθηκε σε ορισμένα από αυτά. Γνωρίζουμε πως η απειλή της τρομοκρατίας σε κάποια κρατημέλη παραμένει εξίσου δυνατή όπως και παλιότερα. Και αν δεν ε, κρυθεί αυτή η προσωρινή συμφωνία, η διάμεση συμφωνία θα είναι ένα μεγάλο χτύπημα στην ασφαλειά μα. Ορισμένοι υποστηρίζουν πω αφού το κάναμε στο παρελθόν, το κάνουμε και στο μέλλον. Μα είπαν πω ε, οι αξιόπιστες πληροφορίε που, δίνουν, ε, που δίνει το TFTP για του γνωστού και ύποπτου τρομοκράτε είναι πολύ σημαντική στήριξη που χρειάζεται ε, που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες απειλές κυρίως από την Αλκάιντα. Αυτή η συμφωνία δεν είναι μόνο υπέρ του, τον ΙΠΑ, είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Πολλά βεβαίως υπόθηκαν για το επίπεδο προστασίας των στοιχείων στην ε, ενδιάμεση συμφωνία και φυσικά αυτό είναι και η ανησυχία κλειδί. Ενθαρρύνω τα μέλη και φαντάζομαι πως όλοι το έχετε κάνει να εξετάσουν πιο στενά αυτή την συμφωνία γιατί θα δείτε ότι περιέχει σημαντικές και λεπτομερείς νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία το Υπουργείο Οικονομικών. τον είπα. Ας πούμε, περιλαμβάνεται αυστηρός περιορισμός για τους στόχους της χρήσης των στοιχείων, δηλαδή έρευνα για την τρομοκρατία. Απαγορεύεται επίσης η, η, εξαγωγή στοιχείων και επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που πιστεύετε πως ο ύποπτος είναι ύποπτος για τρομοκρατία. Αυτό σημαίνει πως τα στοιχεία αυτά είναι ανώνυμα και μόνο αν υπάρχει περίπτωση και πιστεύουμε ότι ένα συγκεκριμένο άνθρωπο θεωρείται ε, ύποπτο τρομοκρατία, μπορούν τα στοιχεία του να βγουν από τη βάση δεδομένων. Επίση, ε, θα πρέπει να διαγράφονται τα στοιχεία εντό των 5 ετών από την παραλαβή του, πράγμα το οποίο συμφωνεί με την ε, σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και εμείς θα συμμετέχουμε στην προστασία των ε, στοιχείων και εμεί θα συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται αυτές οι ε, εγγύησεις. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως μόνο ένα τμήμα των στοιχείων SWIFT θα διαβιβαστούν υπό την διάμεση αυτή συμφωνία και αυτό δεν επηρεάζει τις εξουσίες των αρχών προστασίας των δεδομένων σε σχέση με την διαβίβαση των στοιχείων στις ΕΠΑ ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έχουμε ας πούμε διμερεί σχέσει με, ε, με την Ολλανδία. Οι συγκεκριμένε δικλείδε ασφαλείας δεν θα ισχύουν πλέον. Και αν η ενδιάμεση συμφωνία καταπέσει είναι πολύ πιθανό να περάσει πολύ καιρό πριν ε, μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια εναλλακτική. Άρα λοιπόν η άρνηση της συγκατάθεσης μπορεί να οδηγήσει σε κενό ασφάλειας των δεδομένων και ασφάλεια γενικότερα. Τέλος, Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, η ενδιάμεση αυτή τη συμφωνία είναι μόνο μια προσωρινή συμφωνία. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη του κόσμου, αλλά μπορεί και θα βελτιωθεί. Η Κομισιόν τώρα οριστικοποιεί το σχέδιο εντολή και τι κατευθυντήριε γραμμέ για την μακροπρόθεσμη συμφωνία και θα τα υιοθετήσουμε σύντομα. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι για να διαβεβαιώσω ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πλήρως σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε πως αυτές οι απαντήσεις, πως αυτά που είπα απαντούν σε κάποια από τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για αυτές τις ε, επεξηγήσεις και τη δήλωσή σας που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Πρόκειται για δηλώσεις ε, οι οποίες έγιναν από το Συμβούλιο καταρχήν και έπειτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνδέονται με τι δικέ μας προσδοκίες όσον αφορά το μελλοντικό, μελλοντική διαπραγματευτική εντολή καθώς και την ενημέρωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι πως το Ευρωκοινοβούλιο καθίσταται συνυπεύθυνο για την νομοθεσία στην Ευρώπη. Έχουμε ευθύνε και για τις διεθνείς συμφωνίες ε, τέτοιου τύπου, όπως αυτή που αφορά το SWIFT, ε, θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα και να πούμε πως η κατάσταση μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ πως οι ε, τελευταία μηνύματα από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης δείχνουν πως η κατάσταση αυτή είναι κατανοητή. Το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα έχει πλήρη ευθύνη για την νομοθεσία. Θα θέλαμε αυτό το μήνυμα να είναι ισχυρό και γνωρίζουμε πως είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους πολίτες μας και τους εκλογείς μας. Εμείς εκλεγόμαστε άμεσα ως βουλευτές και έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες μας για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία. Τώρα, ανοίγουμε τη συζήτηση. Εξ του ΕΛΚΑ το λόγο έχει ο κύριος Στράσερ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Πρώτα απ' όλα θέλω στην πρώτη αυτή ημέρα εργασιών να σας καλοχαιρετήσω και εξ ονόματος της ομάδας μας να προσφέρω την καλή και ε, καρποφόρα συνεργασία μας. Θέλουμε και έχουμε μια καλή εταιρική σχέση με τις ίπα ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αυτό πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, είμαστε υπέρ της ασφάλειας των πολιτών σίγουρα και εξίσου είμαστε υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τρίτον, καταβάλαμε προσπάθειες ε, ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου να υπάρξουν οι κατευθυντήριες γραμμές ε, για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων και καθορίσαμε τις θέσεις μας τότε ήδη θέσεις αυτές που τώρα θέλουμε να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν χειροπιαστά. Και τέταρτον, επιτρέψτε μου από πλευρά ε, Επιτροπή, κυρία Επέτροπε, εμεί είμαστε υπεύθυνοι, συνομοθέτε υπεύθυνοι για το νομοθετικό έργο πλέον ως Ευρωβουλή και θέλουμε να συμμετέχουμε ισότιμα με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τώρα, αν δούμε το κείμενο αυτό, δύο πράγματα πρέπει να διαπιστώσουμε. Πρώτον, τον τρόπο πώς απέρευσαν και κατέληξαν αυτά τα κείμενα. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε ως διεργασία, ως διαδικασία. Και δεύτερον, πρέπει να το πω, όταν λέει το Συμβούλιο ελήφθησαν υπόψη σε βάθος τα σημεία από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, κάποια σημεία δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη, πρέπει να πω. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής, διαγραφή στοιχείων κτλ. Αυτοί ήταν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους είπαμε στην Επιτροπή για τα θέματα ασφάλειας ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το κείμενο αυτής της συμφωνίας. Και τώρα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι μόνο μετά από την τοποθέτησή μας κινητοποιήθηκαν κάποια πράγματα. Η Υπουργός Εξωτερικών τον είπα δεν είπε τίποτα άλλο εκτός από το ότι λέει το Συμβούλιο έχει άλλα στοιχεία από εκείνα που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο και αυτή την εβδομάδα δόθηκαν κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα από το Συμβούλιο, αλλά όχι εγγυήσει και χέγγια. Και το λέω αυτό και γι' αυτό για μα το αναφέρω. Θέλω να εξετάσουμε το θέμα περαιτέρω. Θέλουμε μια καλή συμφωνία. Είμαστε απόλυτα υπέρ του να συνεχιστεί η συζήτηση υπέρ αυτών των θεμάτων για να υπάρξει μια καλή συμφωνία. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Θα ήθελα να παρακαλέσω να μην ξεπερνάτε το χρονικό όριο στι παρεμβάσει σα να μην υπερβαίνετε τα χρονικά όρια ως αγορητές. Εντάξει, ο κύριος Μάρτιν Σούλτς παρακαλώ, από πλευράς των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, ο Ιρλανδός συγγραφέας Τζόναθαν Σουίφτ στο βιβλίο του «Τα ταξίδια του Γκιούλιβε» έστειλε τον Γκιούλιβε σε ταξίδι στον κόσμο. Ο Σουίφτ τον έστειλε στη χώρα των Νάνων των Λιλιπούτιων. Ο Γκιούλιβερ όμω ε, ανακάλυψε ότι έφτασε στη χώρα των γιγάντων. Έτσι. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται να συμβαίνει και με την Αμερικανική διπλωματία. Α, ανταποκρίθηκε στις συνήθειες του Γκιούλιβερ. Νόμιζε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νάνο. Όμω φάλμα αυτό από πλευρά τη διπλωματία των ΗΠΑ. Τώρα πρέπει να αναγνωρίσουν Σεσίλια Μάλμστρομ και αυτό με τα συγχαρητήριά μου για την εκλογή σα ω Επιτρόπου περάσατε από το ένα χαρτοφυλάκιο στο άλλο ότι δεν πρόκειται μόνο για σφάλμα τη Αμερικανική διπλωματίας αλλά και τη ε, της κυβέρνησης όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θεώρησαν ότι μπορούν να καταλήξουν με το Ευρωκοινοβούλιο χωρί να αντιληφθούν ότι με μια τόσο ελληματική συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει έγκριση από πλευρά μα. Αυτή η συμφωνία αποπνέει την νοοτροπία της αιμονής για θέματα ασφάλειας όσον αφορά τις ΗΠΑ. Αλλά δεν έχει καθόλου δεν ανταποκρίνεται με το πνεύμα προστασίας των ελευθεριών των πολιτών μας. Πνεύμα το οποίο προέρχεται από την Ευρώπη. Η διαβίβαση μεγάλων όγκων δεδομένων χωρίς εξειδίκευση, χωρίς χειροπιαστά εξειδίκευση σε επιμέρους περιπτώσεις είναι μία θεμελιώδης αντίφαση σε εκείνα που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλίζονται όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και αναγκάσαμε να είναι σεβαστά στην Ευρώπη και στα εθνικά κοινοβούλια. Τα σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την προστασία των ε, δεδομένων αναφέρθηκαν. Επί ποια διάρκεια θα αποθηκεύονται αυτά τα στοιχεία, ποιο θα διαβιβάζει αυτά τα στοιχεία σε ποιον, ποια δυνατότητα έχω να ενημερωθώ εγώ τι συμβαίνει με τα δικά μου προσωπικά δεδομένα, σε ποιον διαβιβάζονται περαιτέρω, αν είναι σωστά αυτά και τι γίνεται και πώς μπορώ να προστατευτώ νομικά, να μην υπάρχουν κάποια εσφαλμένα στοιχεία για μένα που να κατα... Ε, αποθηκεύονται και να διαχετεύονται και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιωτελώς τρίτο. Ποιος μπορεί να διαγράφει αυτά τα στοιχεία, επί ποια διάρκεια θα ε, τηρούνται. Σύμφωνα με το Homeland Security Act, το νομοθέτημα τον είπα για 90 χρόνια Τώρα δεν έχω την εγγύηση ότι θα, γίνω φτάσω τα 90, αλλά μέχρι 90 χρόνια μπορούν να αποθηκεύονται αυτά τα στοιχεία. Όλα αυτά τα σημεία είναι σημαντικές ελλείψεις και ελαττωματικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Για αυτούς τους λόγους κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε ε, Ρουμπαλκάμπα, πρέπει να πω ότι είναι μια κακή συνθήκη αυτή. Καθόλου καλή και δεν μπορούμε να την εγκρίνουμε και απορρίπτοντα την εσείς θα έχετε την εντολή με τη ΣΥΠΑ να ξαναδιαπραγματευτείτε για μια νέα καλύτερη συνθήκη, καλύτερη συμφωνία που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα για την ασφάλεια αλλά και θα διασφαλίζει και τα συμφέροντα των πολιτών μας ε, όσον αφορά τις ελευθερίες τους ε, και τα προσωπικά τους δεδομένα. Είμαστε υπέρ και της ασφάλειας αλλά και της προστασία των δεδομένων. Να εξευρεθεί ένας τέτοιος συμβιβασμός μεταξύ των δύο πρέπει να είναι στόχος των νέων διαπραγματεύσεων. Εγώ δεν μπορώ να συστήσω στην ομάδα μου με αυτή τη μορφή που έχει η συμφωνία να υπερψηφίσει. Θα προτείνω να απορρίψουμε απόψε τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σούλτ η κυρία Σοφή Ιντφέλτ στη συνέχεια, εξ ονόματο τη ομάδα Άλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλωσορίσατε στην καλή μου φίλη και πρώην συνάδελφο Σεσίλια Μάλστρομ. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που εμείς ε, είμαστε υπεύθυνοι ως Κοινοβούλιο και είναι πολύ ψηλές οι προσδοκίες. Αλλά θα πρέπει ε, να, κάνουμε, να λάβουμε μια απόφαση μετά από, πολλές, ε, από πολύ ψύχρεμη διαδικασία. Θα πρέπει να Μην ξεχνάμε, πως είπα, ούτως ή άλλως μπορούν να πάρουν τα στοιχεία χωρίς τη δικιά μας συμφωνία ή διαφωνία. Εμείς μπορούμε μόνο να συγκατατεθούμε σε μια συμφωνία που έχει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα επί τη βάση της ουσίας και της διαδικασίας δεν είναι ένα θέμα μπραντεφέρ ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ούτε αφορά την νομοθεσία μόνο, αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν το, έχουν δικαίωμα για διαφανή και δημοκρατική διαδικασία. Οι απαντήσεις του Συμβουλίου μέχρι στιγμής είναι απαράδεκτες και ακατάλληλες και δεν μπορούμε εμείς να παζαρεύουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών με υποσχέσεις των είπα για μελλοντικέ υποχρεώσει. Το Συμβούλιο είχε αμέτρητε ευκαιρίε από το 2007 να το χειριστεί αυτό σωστά και να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών ε, στοιχείων και των πολιτικών ελευθεριών, εξασφαλίζοντα το δημοκρατικό έλεγχο από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από την 1η Δεκεμβρίου από το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά το, το Συμβούλιο έδειξε μεγάλο πείσμα, απίστευτο πείσμα. Δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση αν δεν έχουμε πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τι πληροφορίε, και οι ψηφοφόροι μα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ότι εξετάζουμε όλα τα στοιχεία πολύ σοβαρά και ότι δεν απλώ σφραγίζουμε, επισφραγίζουμε τι αποφάσει του Συμβουλίου, του Ευρωκοινοβούλου ήταν σαφέ εδώ και χρόνια για τις ανησυχίε του και τις προσδοκίε του. Και αντί να μας δίνει περισσότερες αόριστε υποσχέσεις, το Συμβούλιο θα πρέπει επιτέλου να μας δώσει την άποψη της νομικής του υπηρεσία και τις απαιτούμενε πληροφορίες, δείχνοντας την χρήση των στοιχείων για στόχου αντιτερομοκρατικού και δεν θεωρώ πως η έκθεση αυτή είναι, είναι Αν Άμα θέλετε λοιπόν τη συγκατάθεσή μας θα πρέπει να ανταποκριθείτε στα αιτήματά μας. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος. Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρεμπέκα Χάμς, εξ ονόματος των Πρασίνων. Αυτό ως εκ παρατήρηση σε σχέση με τις επαφές με τους πραγματογνώμονες ε, των ΗΠΑ. Στις δύο αυτές ε, συζητήσεις που είχα δεν αισθάνθηκα καθόλου Ευρωπαία νάνος ή ότι η Ευρώπη είναι νάνος. Το αντίθετο, μέσω αυτών των επαφών με πραγματογνώμονες από τις ΗΠΑ κατάφερα να αποκομίσω πολλά πράγματα και έμαθα πάρα πολλά πράγματα Γιατί τελείως διαφορετικές από πλευρά συστημικής αντιμετώπισης, ε, από πλευρά δομών των θεμάτων ασφάλειας. Και είμαι ευγνώμων στους Αμερικανούς, στη ΣΥΠΑ, ότι από αυτό το διάλογο κατάφεραν να βρουν τους Ευρωπαίους απέναντί τους ως εταίρους για να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να επιτελεστούν. Και το Συμβούλιο δεν το κατάφερε. Δηλαδή να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις ποιε προκλήσει αντιμετωπίζουμε εμεί ω Ευρώπη σε σχέση με την αποτελεσματική καταπολέμηση τη τρομοκρατία αφενό, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ποιε προκλήσει πρέπει να ξεπεράσουμε και είναι πραγματικά έσχο ότι πρέπει να περάσουν τον Ατλαντικό οι Αμερικανοί για να μα καθορίσουν και να επεξηγήσουν αυτό το πεδίο που πρέπει να καλυφθεί, που μέχρι σήμερα δεν κατάφερε το Συμβούλιο να καλύψει στι δράσει του. Η εισηγήτρια κατέστησε απόλυτα σαφές σε ποιου τομεί ε, θεμελιώδη δικαιώματα <clears throat> όπω αυτά τα οποία έχουν μέγιστη προστασία στην Ευρώπη, πώ αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται καθημερινά. Ένα πράγμα θέλω να προσθέσω, που υπό το νομικό πρίσμα και υπό το πολιτικό πρίσμα θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικά πράγματα όταν ασχολείται κανεί με αυτά. Ο ορισμό του τι είναι τρομοκρατία στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη είναι τελείω διαφορετικό από τη μία και άλλη όχθη του Ατλαντικού. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο τίθεται ενώπιον αυτής τη συμφωνία. Κυρίε και κύριοι, σωστά αναφέρθηκε ότι εδώ οι ευρωβουλευτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνοι έναντι των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να λογοδοτούν έναντι των πολιτών για το αν πράγματι μεριμνούν ώστε τα δικαιώματά του να παίρνουν σάρκα και οστά χειροπιαστά και να διασφαλίζονται. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε μια συμφωνία που πολλοί από εμά δημόσια, ο κύριο Βέμπερ, ο κύριο Λάγκ δεν παρίσταται, ο κύριο Σούλτ πάντα εξηγούσαν ότι παραβιάζει ισχύω ενισχύει δίκαιο Πρέπει τώρα να καταφέρουμε, μια και στους πολίτες έναντι της δημόσιας συζήτησης το προαναγγείλαμε, πρέπει να είμαστε ε, υπέρ της ε, ε, συνθήκης αυτής προσωρινής συμφωνίας και όχι υπέρ αναβολής. Δεν επιτρέπεται το Κοινοβούλιο να απεμπολίσει για άλλη μια φορά τις ευθύνες του. Αυτό το κάναμε ήδη τον Νοέμβριο μια φορά. Εκεί θα είχαμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε το χειρόφρενο. Πλειοψηφικά δεν το θελήσαμε τώρα. Τώρα πρέπει να κάνουμε ένα άλμα. Να κάνουμε ένα άλμα και ακριβώς μετά από τις διαβουλεύσεις με τους Αμερικανούς, σας το λέω αυτό, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη θέση, πιο ισότιμη θέση για να μεριμνήσουμε υπέρ της ασφάλειας και υπέρ περισσότερων πολιτικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τίμωθη ε, Κίρκοπ θα λάβει τώρα τον λόγο. Πρόεδρε, όπως και οι υπόλοιποι, Είχα απογοητευτεί και εγώ και θύμωσα πολύ από τη συμπεριφορά του Συμβουλίου ως προς τη διαβούλευση με εμά. Η κοινοβουλευτική διαβούλευση δεν γίνεται εκ των υστέρων. Η αμοιβαιότητα της προστασίας των δεδομένων πρέπει να είναι πλήρης. Και δεν πρέπει να επαναληφθεί τέτοια διαδικασία. Μου έχουν δοθεί βέβαια διασφαλίσεις από τις Αμερικανικές αρχές ο, λόγω των ε, εγγυήσεων που υπάρχουν εκεί ότι θα υπάρξει κάποια προστασία. Δεν πρέπει όμως αυτά να είναι προηγούμενα για μελλοντικές συμφωνίες με τα ΣΥΠΑ. Μας έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Εγώ δεν μπορώ ακόμη να κρίνω αν αυτές οι υποσχέσεις ανταποκρίνονται στις ανησυχίες μας. Χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο πριν προχωρήσουμε με την εξέταση αυτού του σημαντικού μέτρου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λότα Μπίσκι εξ ονόματος της Ενωτικής Ομοσπονδιακής Αριστερά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Συμφωνία SWIFT μέσω μιας αμφισβητήσιμης διαδικασίας αντιμετωπίστηκε και καλύφθηκε και πολύ γοργά, ακόμα μία μέρα κιόλα πριν από την έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα, ε, ε, υλοποιήθηκε, επικυρώθηκε ώστε να παρακαμφθεί το Κοινοβούλιο. Εγώ κυρίω θέλω να επικεντρωθώ στην ουσία. Εδώ έχουμε δίπλα στον κοντά στον μεγάλο αδερφό Big Brother, Little Sister, τη μικρή αδερφή. Πιστεύει η κυρία Χίλαρη Κλίντον ότι μπορεί να μας πείσει εμάς ερετούς ευρωβουλευτές αυτό το οποίο εμείς δεν δεχόμαστε από τις κυβερνήσεις μας. Δηλαδή είναι απόλυτα λανθασμένο ε, τα, θέματα τρομοκρατίας ε, να αντιμετωπίζονται με τέτοια ευρεία παρέμβαση σε τράπεζες δεδομένων προσωπικών, δικαιωμάτων, ε, προσωπικών δεδομένων. Διότι έτσι η αξιοπιστία μας υπονομεύεται. Επί δεκαετίες αποθηκευόντουσαν τέτοια προσωπικά δεδομένα χωρίς κανένα έλεγχο. Ούτε και καν για την περίοδο, για τη διάρκεια της αποθήκευσης. Και όσον αφορά επίσης και την αποζημίωση λόγω εσφαλμένης χρήσης δεν μπορεί κανείς να ασκήσει προσφυγή. Εδώ έχουν, έχουν οι κυβερνήσει τα κράτη προτεραιότητα εναντί των πολιτών και υποβαθμίζονται οι πολίτες σε υπόπτους συλλήβδην. Μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις ακολουθούν μια πολιτική παρακολούθηση των πολιτών. Για να έρθω στο γερμανικό παράδειγμα, η Telekom, η Deutsche Bahn, η λόγω των πρακτικών εκεί θα πρέπει, δεν θα πρέπει να ισχύνονται, να ντρέπονται για την συλλογή στοιχείων και την παρακολούθηση των εργαζομένων τους. Τώρα στοιχεία αγοράζει η γερμανική κυβέρνηση όσον αφορά καταθέτες που έχουν καταθέσει στο εξωτερικό και συλλέγουν στοιχεία εις βάρος τους. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου εμείς ως βουλευτές πρέπει να λάβουμε απόφαση επ' αυτών. Γιατί το Google θα ε, έχει ε, αναπτύσει, αναπτύσει αυτές τις πολιτικές από πλευράς του. Η τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί κυρίως τα αίτια, οι ρίζες της τρομοκρατίας. τρομοκρατίας. Εκεί συμφωνούμε όλοι. Αλλά όχι ε, υπονομεύοντας ή απεμπολώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα. Μια από αυτές τις αξίες ακριβώς με το SWIFT είναι εκείνο το οποίο απεμπολούμε και αγνοούμε. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να δεχθεί όμω η ομάδα μου. Θα καταψηφίσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακολουθήσουν οι άλλοι εγγεγραμμένοι αγορητέ, ο κύριο Μπουσουτή. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι το ΕΛΚ είναι υπέρ τη συμφωνία αυτή, υπέρ τη συμφωνία SWIFT δηλαδή, και αύριο θα υπερψηφίσει. Θα σας εξηγήσω όμως γιατί. Είμαστε υπέρ διότι σκεφτόμαστε καταρχάς την ασφάλεια των πολιτών μας. Και η ασφάλεια αυτή θα διασφαλιστεί καλύτερα μετά από την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και εμπειρογνώμονες που ερεύνησαν τα πράγματα ως προς την ασφάλεια στις χώρες που εκπροσωπούμε εδώ. Η ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών μας σίγουρα θα βελτιωθεί με την, με την συμφωνία αυτή. Ακόμα και η ασφάλεια των ΗΠΑ θα βελτιωθεί. Συμφωνώ όμως, όμως ότι το Συμβούλιο δεν έχει φερθεί όπως θα έπρεπε στο, προς το Κοινοβούλιο. Γιατί υπάρχει και μια έκθεση που στάλθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το θέμα της συμπεριφορά του Συμβουλίου και κατανοώ τις ανησυχίες των συναδέλφων για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η συμφωνία αυτή είναι ενδιάμεση προσωρινή που μας επιτρέπει απλώς να προετοιμάσουμε την μόνιμη, τη μελλοντική μόνιμη συμφωνία. Επίσης αναφέρθηκε πρόεδρε το θέμα γενικότερα της ασφάλειας και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να επωφεληθούν από τις νέες μας δικαιοδοσίες για να αντιμετωπίσουμε τα 500 εκατομμύρια πολιτών με ε, την βεβαιότητα να μπορούμε να τους πούμε με βεβαιότητα ότι αγωνιζόμαστε για την ασφάλειά τους. Και για αύριο σας εξήγησα πώς θα ψηφίσουμε. Thank you, President. Uh, we too in the and Democrats want to fight for the European Σας ευχαριστώ. Οι σοσιαλδημοκράτες θέλουμε να υπερασπιστούμε τους Ευρωπαίους πολίτες και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και γι' αυτό και συστήνουμε να ψηφίσουμε όχι αύριο, όπως είπε και ο αρχηγός μας, ώστε να διασφαλίσουμε πως αυτή η διαδικασία ε, κατά μιας, θα είναι μάλλον κατά ε, μάλλον δεν γίνεται σύμφωνα με τη Λισαβόνα, αλλά είναι μια κακή διαδικασία. Το θέμα είναι αν μια συμφωνία που έχει συνταχθεί άσχημα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ασφαλείας και της αντιτρομοκρατίας. Ένας από τους συμβούλους μου, ο κύριος Κέρκοπ είναι δικηγόρος και ο κύριος Κέρκοπ είναι δικηγόρος και είχε πει μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα πρέπει να βάλει την ασφάλεια τόσο, μακριά, τόσο πολύ μακριά ώστε να στερήσει και την ελευθερία. Είναι οπωσδήποτε ε, αλήθεια πως το Συμβούλιο αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα τα οποία και εμείς θεωρούσαμε σημαντικά και μάλιστα αναγνωρίστηκε πως το Κοινοβούλιο είχε εδώ ε, δίκιο γιατί κανένα από αυτά τα κείμενα δεν μας, έδωσαν, ε, δεν μας έδωσε ένα πρόγραμμα για να ε, λύσουμε το πρόβλημα και άλλα, ένα όχι θα μας οδηγήσει μια καλύτερη συμφωνία για ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Η ομάδα μας ε, κάνει έκκληση σε ολόκληρο το σώμα να στηρίξει την εισηγήτρια και αυτό προσπαθεί να κάνει. Δηλαδή, καλύτερη συμφωνία κατά της τρομοκρατίας. Καλύτερη συμφωνία χρειαζόμαστε λοιπόν και αυτό θα συστήσουμε ε, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες απόψε στην ομάδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Δία παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, απορρίπτω τις μεθόδους και τις προθεσμίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμφωνία που συζητάμε σήμερα. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι θεμελιώδους σημασίας και η συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να είναι σεβαστά από όλους η μεγαλύτερη βλάβη που μπορεί να, πάθει, που μπορεί να κάνει μια δημοκρατική κοινωνία στην τρομοκρατία είναι να κόψει την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Γι' αυτό πρέπει η τελική συμφωνία κατεπηγόντως να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το SWIFT και το TFTP έδειξαν την αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση τρομοκρατικών δράσεων και στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική. Ο θεμελιώδης στόχος είναι η προστασία των δεδομένων ποιον ρόλο θα έχουμε του επόπτη ή του ειδικού ε, δικαστή με τις αντιφάσεις που υπάρχουν. Όχι, σε αυτό το θέμα ούτε καν συζητήθηκε, ούτε επετεύχθη μια ε, λύση, μια ενιαία λύση. Είναι ε, η συμφωνία αυτή, η ενδιάμεση συμφωνία λέει ότι τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή τρομοκρατικών πράξεων. Δεν θα συνδέονται με άλλες βάσεις δεδομένων. Θα έχουν μόνο πρόσβαση τα σώματα ασφαλείας. Εμπιστεύομαι την κυβέρνηση των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε την υποχρέωση να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ ως φυσικό εταίρο απέναντί μας. Για όλους αυτούς τους λόγους υποστηρίζω να την προσωρινή συμφωνία αυτή και πρέπει να υπερψηφίσουμε ως Ευρωβουλή και να αναγνωριστούν αυτά από πλευρά τον είπα και από πλευρά Χίλαρη Κλίντον και Γκέιτνερ. Εν τέλει, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να τηρήσουν. Είναι κατεπήγον να υπάρξει μια διοργανική συμφωνία. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο παρακαλώ για ένα Κύριε Πρόεδρε, μια απλή επιστολή του Συμβουλίου ότι οι διαπραγματεύτικέ γραμμέ θα συμπεριλαμβάνουν τι ανησυχίε του Κοινοβουλίου θα σημαίνει ότι αρχίζουν αμέσω οι διαπραγματεύσει με τις ΥΠΑ, όχι κάποτε στο μέλλον, αλλά αμέσω. Εάν υπάρξει υπόσχεση ότι θα παίξει το ρόλο του το Κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να αρκέσει και θα καθησύχαζε έτσι όλους τους συναδέλφους που έχουν θεμητές ανησυχίες. Και σήμερα μπορεί να γίνει αυτή η επιστολή. Ο Επίτροπος είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η καθεαυτή μεταφορά των δεδομένων. Υπάρχει το SWIFT. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επίσης μας διασφαλίζουν ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αναφέρατε ότι οι διαπραγματευτικές γραμμές έχουν περίπου συμφωνηθεί. Πού είναι όμως. Αφού έχετε αυτή την πίεση σήμερα, γιατί δεν μας λέτε πού συμφωνείτε και πού διαφωνείτε με το Κοινοβούλιο ακριβώς αντί για γενικές δηλώσεις. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε μαζί με τη ΣΥΠΑ την τρομοκρατία και γι' αυτό ζητώ και από το Συμβούλιο και από τη ΣΥΠΑ να συνεργαστούν σοβαρά μαζί μας μετά την αυριανή ψηφοφορία, όχι χωριστά ο καθένας ούτε να ονειρεύονται ότι θα καταστρέψουν την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Παρακαλώ συνάδελφοι να μην μιλάτε παραπάνω από ό,τι προβλέπετε. Ο κύριος Ζέμκε. Ζέμκε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο όμως είχα ζητήσει τον λόγο για να παρέμβω στη διαδικασία Catch the Eye, εντάξει. Ε, ε, πάνη Birgit Zippel. Birgit Zippel παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος τις πολλές συζητήσεις ε, για το SWIFT τις τελευταίες εβδομάδες τις έχει παρακολουθήσει θα μπορούσε να αποκομίσει την εντύπωση χωρίς το SWIFT ε, θα επέλθει το χάος. Μια απόρριψη αυτής της συμφωνίας θα διακόψει πλέον, θα τερματίσει τις διατλαντικές ε, σχέσεις και θα διακόψει και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτές οι απειλές μπορούν να ε, χαρακτηριστούν με μία λέξη. Είναι γελίες. Οι ε, ΙΠΑ ε, κάνουν την προσπάθεια να σώσουν τα προσχήματα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός συμφωνιών και μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το SWIFT θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο λιθαράκι η αποτυχημένη προσπάθεια της 25ης 12ης δείχνει ότι δεν λείπουν τα στοιχεία χρειάζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των στοιχείων. Η ενδιάμεση συμφωνία είναι πολύ κακή, πολύ αρνητική. Είναι αντιφατική. Αντί να βρίσκει τις σωστές διεργασίες ώστε μόνο στοιχεία πραγματικά υπόπτων να διαβιβάζονται και να ανταλλάσσονται, συλλήβδιν ανταλλάσσονται στοιχεία με τη ΣΥΠΑ που πραγματικά τα πολιτικά δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων τα παραβιάζουν. Και τώρα αν οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες ε, να εισακούσουν μια τέτοια, ε, αυτές τις επικρίσεις ε, και να καταλήγαμε σε μια καλή συμφωνία δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να έχει εγκριθεί αυτή η αρνητική συμφωνία. Θα πρέπει να ισχύει το όχι κατά της προσωρινής συμφωνίας. Να αρχίσουν άμεσες νέες διαπραγματεύσεις ώστε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια θετική συμφωνία. Να έχουμε ένα αποτελεσματικό μέσο στα χέρια μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προστασία των πολιτών μας. Ο κύριος Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγγιλάρ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας άνοιξε μια νέα περίοδο για αυτή την Ευρωβουλή, αλλά επίσης και για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παρέμβαση του Υπουργού Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, κ. Ρομπακάμπα, σημειώνει ότι αυτή η Ευρωβουλή πρέπει να εισακούγεται και τα αιτήματα και οι απαιτήσει και οι διεκδικήσει πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Δεύτερον, σημειώνει ότι η διαπραγμάτευση αυτή τη συμφωνία δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο, δεν έγινε επαρκώ με καλό τρόπο, αλλά κυρίω δεσμεύτηκε εναντί του μέλλοντο και είπε θα διαπραγματευτεί το δυνατόν γοργότερα μια τελική καθοριστική συμφωνία ώστε να καλυφθούν τα αιτήματα τα οποία εκφράζονται από την έκθεση της εισηγήτριας αιτήματα εχέγγυων, πρόσβασης και άσκησης προσφυγής και δικαίωμα γνωστοποίησης ή και διαγραφής όσον αφορά στοιχεία προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να εξευρεθεί μια νέα ισορροπία μεταξύ της διαφύλαξης της προσωπικής ζωής, των στοιχείων των πολιτών και των δικαιωμάτων των πολιτών που εκπροσωπούμε εμείς στην Ευρωβουλή. Οποιοδήποτε και να είναι το αποτέλεσμα στη συζήτηση ενθαρρύνει και προτρέπει κύριε Υπουργέ το δυνατόν να μπορέσετε να προχωρήσετε σε αυτέ τι διαπραγματεύσει για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σε σχέση με συνθήκε τη Λισαβόνα, τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την εκπροσώπηση 500 εκατομμυρίων πολιτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Διαδικασία catch the eye τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ εσείς, κύριε λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ χωρίς ε, μια πραγματική αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων στην περίοδο της κινητικότητας δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια. Έχουμε κάθε λόγο τους πολίτες μας να τους προστατεύουμε έναντι τρομοκρατικών αποπειρών και πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της διαφύλαξης της προσωπικής ζωής και προσωπικών στοιχείων των πολιτών μας. Και μια τέτοια ισορροπία πρέπει να εξευρεθεί σε αυτή τη συμφωνία δεδομένων όλων αυτών των θεμάτων. Αν αυτό είναι τόσο σημαντικό, τότε η στάση του Συμβουλίου ήταν ερασιτεχνική μέχρι τώρα και παρακαλώ να υπάρξουν περισσότερα, περισσότερες δεσμεύσεις όσον αφορά την εισηγήτρια ώστε ίσως έτσι να μπορέσουμε να καταφέρουμε να επιτύχουμε πλειοψηφία υπέρ αυτής της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο. Εφόσον δεν έχουμε αυτά τα εχέγγυα, το πρόγραμμα TFTP, εφόσον δεν έχουμε όλα αυτά τα εχέγγυα, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί το SWIFT να παίρνει εξειδικευμένα στοιχεία. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η εγγύηση και όλα αυτά δεν επιτυγχάνονται, αυτή η συμφωνία είναι σημαντική και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να οδεύσουμε προς την αναβολή και τέλος τέλος με αυτόν τον τρόπο να ρυθμίσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντική η συζήτηση. Δεν θέλω να σας αρχίσω να σας διακόπτω, αλλά βλέπετε ότι όλοι σας ε, μακρηγορείτε μισό λεπτό παραπάνω. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε 11 ανθρώπους στον κατάλογο. Άμα μιλάτε τόση ώρα, δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους. Επόμενος είναι ο κύριος Λάιχτφριτ. Λάιχτφριτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κανείς δεν αμφιβάλλει σοβαρά για την ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Όμως, η, στη δημοκρατία το κράτος δικαίου πάντα είναι το θέμα πώς γίνεται, πώς ε, επιτυγχάνεται κάτι, με ποιο τρόπο και ποιες διεργασίες. Και εδώ είναι πολύ απλό να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Όχι έτσι όπως τα 500 εκατομμύρια άτομα πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όχι με το να καθίστανται ύποπτοι αυτοί οι πολίτες χωρίς να έχουν δυνατότητα να προστατευθούν και κυρίως όχι με τον τρόπο αυτό, αυτών των μέτρων με περιφρόνηση των ε, δημοκρατικών ρυθμίσεων. Και τώρα Εμεί εμείς εδώ ως Κοινοβούλιο πρέπει να δεχθούμε όλα αυτά που η αλαζονία της Προεδρίας του Συμβουλίου έδωσαν ως αποτέλεσμα στο παρελθόν. Όχι, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Είναι απαράδεκτο και γι' αυτό είμαι υπέρ αύριο να καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Κύριε Λάιχτφριτ, ο κύριος Σλούτερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω πως μπορούμε να ψηφίσουμε εγκρίνοντας αυτή την έκθεση. Εδώ αναφέρατε τέσσερις επιθέσεις τρομοκρατικές που δεν παρεμποδίστηκαν λόγω χάρη μάλλον στις υπησχύουσες συμφωνίες. Λείπει η ασφάλεια λοιπόν. Με αυτήν την συμφωνία υποτίθεται ότι μπορεί να υπάρξει ένα σύστημα επαγρύπνησης ακόμα και με το σύστημα Big Brother δεν μπορούμε να αποφύγουμε να γίνονται επιθέσεις είτε στο ίντερνετ είτε στον ε, τραπεζικό τομέα οι τρομοκράτες ε, πάντα θα βρίσκουν τρόπους για να επιτίθενται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει διαρκής και άμεση επαγρύγνηση. Τι σημαίνει αυτό ε, όταν είναι εις βάρος της ακεραιότητας, της ελευθερίας και της ιδιωτικής ζωής των συμπολιτών μας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να δουλεύουμε με έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί και κλεισμένο το θυρών. No, resign. Παν Κοχ. Παν Κοχ. Κοχ παρακαλώ. Για το επόμενο θέμα ήθελα να παρέμβω, όχι αυτό. Παν Ζέμκε. Ζέμκε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επισύρω την προσοχή σας σε δύο σημαντικά θέματα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία, σίγουρα. Όμως η συζήτηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και ποια συμφωνία θα υπογραφεί ή θα υπογράφαμε με τη ΣΥΠΑ. Έχω δύο παρατηρήσεις ε, στα εξής θέματα. Πρώτον, αυτή η συμφωνία είναι πολύ μονομερής. Είναι μονοβαρής, μονο, μονόπλευρη συμφωνία. Προβληματιστήκαμε καθόλου και είδαμε ότι οι αντίστοιχε υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών μελών θα, θα έπρεπε να μπορούν να αντλήσουν στοιχεία από τη ΣΥΠΑ που θα ήταν ίσως χρήσιμα για μας στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεύτερο, η κυριότερη επιφύλαξη αφορά το γεγονός ότι όλα τα δεδομένα χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όλα αυτά τα δεδομένα θα μπορούν να αντλούνται. Θα πρέπει όμως να μπορέσουμε να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι μυστικές υπηρεσίες των ΙΠΑ και της ΕΕ αποκλειστικά τα στοιχεία των υπόπτων θα έπρεπε να αντλούν και όχι όλων των πολιτών. Κύριε Μαρινέσκου, παρακαλώ έχετε τον λόγο. Consiliul a trimis acordul către Parlamentul European foarte târziu. Σα ευχαριστώ. Το Συμβούλιο καθυστέρησε και γνωστοποίησε στο Κοινοβούλιο με μεγάλη καθυστέρηση τη θέση του. Αυτό ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον γιατί είναι απαράδεκτο. Από την άλλη πλευρά, ευχάριστα εξεπλάγει για τη συνεργασία των αρχών των ΗΠΑ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτή η θετική συνεργασία. Το ίδιο, ε, με το ίδιο ε, το ίδιο ενδιαφέρον αναμένουμε να καταδείξουν οι ΙΠΑ όσον αφορά το πρόγραμμα Visa Waiver, δηλαδή απαλλαγή χορηγήσεων θεωρήσεων διαβατηρίων για υπηκό των ε, ευρωπαϊκών κρατών μελών. Αρνούνται, είπα, να ε, καλυφθούν ε, κάποιες χώρες, οι πολίτες κάποιων χωρών από αυτή την απαλλαγή. Παρ' όλα αυτά όμως η ανταλλαγή των στοιχείων SWIFT είναι σημαντικό στοιχείο για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Δεν θα έπρεπε όμως να γίνονται τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε οι διαπραγματεύσεις τώρα να διακοπούν όταν θα μπορούσαμε να είχαμε και ένα μακροπρόθεσμο ε, τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Κάποιες διαπιστώσεις πρώτα. Το Συμβούλιο ομολόγησε σήμερα ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ίσως δεν είναι το καλύτερο. Θα πρέπει αυτό να λάβουμε υπόψη και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο λοιπόν στο μέλλον. Όμω γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αναβολή. Με αυτή την αναβολή, αυτή, αυτή θα γίνει αναβολή χωρί όρου και προποθέσει. Θα ξαναβρεθούμε στην Ολομέλεια στο μέλλον μπροστά από την ίδια κατάσταση. Δεν θα αλλάξει τίποτα με την αναβολή. Δεύτερον, υποσχέσει ότι θα βελτιωθούν λέει τα πράγματα στο δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων. Χωρί συμμετοχή του Κοινοβουλίου φτάνει πια. Και μα είχαν υποσχεθεί και ήδη με αυτή τη συμφωνία ότι όλα λέει θα γινόντουσαν με διαφορετικό τρόπο και δεν έγιναν. Και πάλι εδώ, όχι αναβολή, δεν βοηθάει εδώ. Μόνο ένα σαφές μήνυμα βοηθάει. Και τρίτο στοιχείο, η, ε, τα κενά για την ασφάλεια, όπου επανειλημμένα αναφέρθηκε ότι θα υπήρχαν αν αυτή την ε, προσωρινή συμφωνία δεν θα την εγκρίναμε, δεν υπάρχουν τέτοια κενά για την ασφάλεια. Και αυτό το λένε όλα ε, οι πραγματογνωμοσύνες που έχουμε στα χέρια μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ασφάλεια των πολιτών μας είναι βέβαια τεράστιου ενδιαφέροντος για όλους μας. Αλλά θα ήταν πολύ εύκολο να μας κατηγορήσουν ότι δεν τηρούμε στεναρή στάση κατά πολέμηση της τρομοκρατίας επειδή ζητούμε την προστασία των πολιτών. Έχει γίνει, έχει ασκηθεί αυτή η κατηγορία πολλές φορές από εθνικούς βουλευτές όταν κρίνουν τη δράση των ευρωβουλευτών. Εμείς υποστηρίζουμε τα παραδείγματα καλής λειτουργίας του SWIFT, αλλά επίσης σωστό θα ήταν να δούμε και τις περιπτώσεις αποτυχιών του SWIFT. Υπήρξαν πολλές αποτυχίες του SWIFT μέσα στην Ένωση και στη δική μου μόνο εκλογική περιφέρεια 12 αθώοι άνθρωποι κρατήθηκαν και χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία γιατί τους ε, είχαν πει ότι οι δοσοληψίες τους ήταν ύποπτες. Τι μας μαθαίνει αυτό, Συμβούλιο, κρατήστε κάποια απόσταση, δεν ε, υφίσταστε πίεση χρόνου, δέστε τα πράγματα ψυχρότερα. Και αυτό δεν το ζητώ μόνο εξ ονόματος των Ευρωβουλευτών, αλλά και των πολιτών όλων. Ευχαριστώ πολύ Κοέλιο. Κύριος Κοέλιο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε στη χώρα μας όταν ένας αστυνομικός που έχει για πρόσβαση σε ένα λογαριασμό χρειάζεται δικαστική εντολή. Δεν μπορώ να δεχθώ μια συμφωνία όπου χιλιάδες ή εκατομμύρια τέτοια στοιχεία θα μπορούν χωρίς τέτοια εντολή να διαβιβάζονται για να εξεταστούν από ένα Αμερικανό αστυνόμο. Υπάρχει έλλειμμα λοιπόν εδώ σε σχέση με αυτή την προστασία των στοιχείων. Δεν είναι πολυτέλεια η προστασία των στοιχείων. Είναι όρος και προϋπόθεσης της ελευθερίας μας. Υπάρχει έλλειψη εδώ ανα και αποτελεσματικότητα. και δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό. Σίγουρα η τελική συμφωνία ελπίζουμε ότι θα είναι μια συμφωνία που θα διαπραγματευτούμε με καλό τρόπο. Πώ θα διαπραγματευτούμε με καλό τρόπο, εκκινώντα από μια αρνητική βάση ή όχι. Είναι καλύτερο να έχουμε μια κακή προσωρινή συμφωνία από το να μην υπάρχει καμιά συμφωνία. Μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση λοιπόν αυτή η προσωρινή συμφωνία για μια καλύτερη τελική συμφωνία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση από πλευράς της κυρίας Βλασσικόβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι το θέμα μιας καλή συμφωνίας. Μια καλή συμφωνία πρέπει να συνάπτεται από ισότιμους εταίρου. Η κατάσταση όμως δείχνει ότι δεν είμαστε ισότιμοι εταίροι εμείς εναντί των ΗΠΑ. Δείχνει μάλλον ότι οι ΗΠΑ απαιτούν κάτι και προσδοκούν κάτι από εμάς και τι προσδοκούν και αναμένουν ότι εμείς θα επαναχωρήσουμε και θα ανταποκριθούμε στα αιτήματα, στα αιτήματά τους και τι απαιτήσει του. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλά περισσότερα δικαιώματα και αρμοδιότητε σύμφωνα με τι συνθήκε τη Λισαβόνα. Θέλουμε και πρέπει τα δικαιώματα των 500 εκατομμυρίων πολιτών τη Ένωση να τα προασπίσουμε και να τα υπερασπιστούμε σωστά. Γι' αυτό είμαι υπέρ τη ε, ε, αναθεώρηση αυτή τη συμφωνία, τη ε, κάλυψη των δικών μα ετοιμάτων, διότι εμεί είμαστε οι μόνοι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένουμε όλα αυτά στην τελική συνθήκη να αντανακλώνται. Ευχαριστώ. Και επίση να προσθέσω ότι πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολλά προβλήματα με την τρομοκρατία. Η Ισπανία έχει μακροπρόθεσμα πρόβλημα με την τρομοκρατία, την οποία καταπολεμά επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε το Συμβούλιο να είναι εταίρο του Κοινοβουλίου. Συνάδελφοι, σας έδωσα δέκα δυνατότητες, δέκα ε, φορές το λόγο, σύμφωνα με το ΚΑΣΔΙΑ και τώρα στρέφουμε στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Κύριε Προεδρεύοντα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να πω και να εκφράσω ότι άκουσα όλους τους ευρωβουλευτές με μεγάλο ενδιαφέρον και ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις εκείνες που υποστήριξαν εμάς και εκείνες που ήταν λιγότερο ε, υποστηρικτικές και τις επικριτικές ακόμα. Ευχαριστώ και για τις επικρίσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω επισημένοντας ότι ευχαριστώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για το ότι διαπιστώνω για άλλη μια φορά σε αυτή τη συζήτηση στην Ευρωβουλή ότι υπάρχει σύμπτωση απόψεων, απόλυτη σύμπτωση απόψεων μεταξύ Ευρωβουλής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου όταν έρχεται η ώρα να προασπίσουμε τις αξίες μας και να αντιμετωπίσουμε με κάθε σθένος την τρομοκρατία. Όπως είπα και στην παρέμβασή μου, αντιμετωπίζοντας οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας. Αυτή είναι η πρώτη συνένεση που πρέπει να υπάρχει ως αναγκαίος όρος. Τώρα, όσον αφορά την συμφωνία που εξετάσαμε απόψε, τη συμφωνία για το SWIFT, θα ήθελα να διαφοροποιήσω μεταξύ των επικρίσεων που έγιναν υπήρξαν δύο μορφές διαφορετικών τοποθετήσεων. Οι επικρίσεις για την μορφή και το, ε, ε, τον τύπο και οι επικρίσεις επί της ουσίας αληθεύει ότι ήταν πιο σταθερέ οι επικρίσει επί τη ουσία και από εκείνου του ευρωβουλευτέ που υποστήριξαν ρητά την ύπαρξη μια συμφωνία σαν αυτήν την συμφωνία που συζητούμε για αυτήν απόψε. Όπω είπα στην αρχική μου παρέμβαση και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι πιθανόν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει με καλύτερο τρόπο από πλευρά του Συμβουλίου. Είναι σίγουρο ίσω ότι μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα. Όμω το είπα και άλλη μια φορά και το επαναλαμβάνω ότι οι προθεσμίε και οι διορίες ήταν πιεστικές και ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε μέσα σε πολύ πιεστικό χρονικό διάστημα να εργαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Εν πάση περιπτώσει θέλω να καταστεί απόλυτα σαφές ότι η βούληση του Συμβουλίου, Συμβουλίου που εκφράζω εδώ απόψε είναι τα πράγματα να μην γίνουν με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον, να γίνουν διαφορετικά με καλύτερο τρόπο. Υπήρξαν κάποιοι ευρωβουλευτές που αμφισβήτησαν Ίσως θα έχουν τους λόγους τους βέβαια για το ότι αυτό ο συμβιβασμός, ε, η υπόσχεση που δόθηκε για ένα συμβιβασμό που δεν τηρήθηκε η υπόσχεση κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι από πλευρά του Συμβουλίου είναι μια δέσμευση που όπως είπα γεννάται από μια δέσμευση επί της ουσίας με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι η συνθήκη της Λισαβόνας που καθορίζει ως θεμελιώδη στόχο η Ευρωβουλή να διαδραματίζει κάθε φορά ένα πιο σημαντικό ρόλο στη θεσμική ζωή τη Ευρώπη, ώστε οι πολίτε αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται καλύτερα. Αυτή είναι η δέσμευση τη Ισπανία, τη χώρα μου, επί τη ουσία. Βαθιά δέσμευση για τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και αυτό με κάνει να πω κατηγορηματικά εδώ ότι το Συμβούλιο, η Ισπανική Προεδρία, θα κάνει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, προσπαθώντα να επιτύχει καλύτερα, καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν κάποιο θέλει να αμφισβητήσει αυτό, είναι δικαίωμά του. Όμω, η συνθήκη υποχρεώνει να κάνουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Αν δεν αρκεί λοιπόν η πολιτική βούληση του Συμβουλίου, υπάρχει η συνθήκη που είναι ο νόμο, ώστε θα διασφαλίσετε ότι τα πράγματα στο μέλλον θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ευελπιστούμε ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το πνεύμα που προασπίστηκε από κοινού από όλου του Ευρωβουλευτέ, ένα πνεύμα που αναζητεί μια ισορροπία μεταξύ τη προάσπιση ασφάλεια και τη διαστήριση διαφύλαξη των αξιών μα, είναι μια δέσμευση που απόλυτα αντανακλάται και στο Συμβούλιο. Για την ίδια την ουσία αυτού του θέματο. Τρία σχόλια θα κάνω. Δεν θα επισέλθω σε πιο συγκεκριμένες πτυχές που αποτέλεσαν αντικείμενο επικρίσεων. Αληθεύει ότι κάποιες από αυτές τις πτυχές ήταν επικριτικές και πολλές φορές ε, δεν ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες. Για παράδειγμα αναφέρθηκε αρκετές φορές ότι η συμφωνία SWIFT όπως ε, έχει αυτή τη στιγμή επιτρέπει χίδιν, σιλίδιν μεταφορά στοιχείων. Και θα έπρεπε να είναι σαφές ότι δεν είναι αυτή η λογική που εμπνέει αυτή τη συμφωνία. Αυτή η χίδιν σιλίδιν συμφωνία μόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπεται από συμφωνία SWIFT και μόνο όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες ε, υποψίες. Στο άρθρο 4 αναφέρεται αυτή η συμφωνία σε αυτό. Τούτου λεχθέντος υπάρχει και μια άλλη σειρά κατηγοριών ή επικρίσεων που έγιναν που νομίζω ανταποκρίνονται μάλλον επιφανειακά στην ουσία της συμφωνίας και έτσι δεν θα απαντήσω σε αυτές τις τοποθετήσεις αυτή τη στιγμή. Επί της ουσίας όμως δύο πράγματα ακόμα θα θέλω να πω. Πρώτον, Εμένω και επιμένω, όπως έκανε και η Επίτροπος πιο πριν, όπως και κάποιοι από εσά κύριε Ευρωβουλευτές, στο ότι αυτό το σώμα όπως είπε, αυτή η συμφωνία πρέπει να είναι χρήσιμη και θα είναι ε, χρήσιμη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έδωσα κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν κάποια άλλα παραδείγματα στην έκθεση του δικαστή που έχουν στη διάθεσή τους οι βουλευτές. Ακόμα ένα παράδειγμα θα δώσω που αναφέρεται στη χώρα μου ή καλύτερα δύο. Αληθεύει ότι η συμφωνία SWIFT χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστούν, να ε, ε, ανοιχνευτούν οι τρομοκρατικές απόπειρες του Μαρτίου, 11 Μαρτίου στην Ισπανία καθώς επίσης και σε σχέση και με την ε, Βαρκελόνη πριν από ένα χρόνο περίπου. Σήμερα όσοι προσπάθησαν να κάνουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις δράσεις βρίσκονται σε ισπανικές φυλακές. Μάλιστα, λειτουργήσε η συμφωνία αυτή και έδωσε αποτελέσματα χειροπιαστά. Και αν συμβαίνει αυτό, τότε θα συμφωνήσετε μαζί μου, κυρίε και κύριοι, ότι αν διακοπεί αυτή η συμφωνία, τότε οι Ευρωπαίοι πολίτε θα ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους και λιγότερο ασφαλείς. Αν λειτουργήσε λοιπόν αυτή η συμφωνία και αν τώρα διακοπεί θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι με αυτή τη διακοπή θα μέναμε λιγότερο ασφαλείς. Χρησιμοποιώ αυτή τη διατύπωση εσκεμένα για να μην μπορεί κανεί να κατηγορήσει το Συμβούλιο ότι δραματοποιεί πράγματα. Θα είμαστε λιγότερο, κάπως λιγότερο ασφαλείς. Γι' αυτό εμένω και επιμένω και ότι ένα, και ένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τη η συμφωνία δεν πρέπει να διακοπεί. Εμένω και επιμένω για άλλη μια φορά. Αυτή η συμφωνία μπορεί να δεχθεί κριτικέ και επικρίσει. Ακούστηκαν σκληρέ επικριτικέ παρατηρήσει απόψε. Αλλά θα συμφωνήσετε μαζί μου κυρίε και κύριοι ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ καλύτερη από το πρωτόκολλο που επί πολλά χρόνια διασφα... κάλυπτε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ. Είναι πιθανόν αυτή η συμφωνία που συζητούμε και εξετάζουμε σήμερα να μην είναι η καλύτερη. Σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί. Και συμπίπτω και συμφωνώ με κάποιε από τι επικρίσει που έγιναν από του Ευρωβουλευτέ. Αλλά να αναγνωρίσετε όμω μαζί μου ότι είναι καλύτερη αυτή η προσωρινή συμφωνία από εκείνο το πρωτόκολλο που υπήρχε πριν. Και έτσι υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί για αυτά τα θέματα που ανησυχούν τους ευρωβουλευτές και που ουσιαστικά στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια δεν θα αποβαίνει εις βάρος ε, των ελευθεριών. Η ασφάλεια δεν θα αποβαίνει εις βάρος των πολιτικών ελευθεριών. Γι' αυτό εμένω και επιμένω ότι είναι σημαντικό, όπως είπε η Επίτροπος, να μην διακοπεί αυτή η συμφωνία, να μπορέσει να λειτουργήσει. Επαναλαμβάνω ενώπιον του Κοινοβουλίου τη βούληση του Συμβουλίου να διαπραγματευτούμε μια νέα συμφωνία. Τελεσίδη και καθοριστική. Μια νέα συμφωνία, στην οποία θα μπορέσουν να ενταχθούν πολλά από τα πράγματα που ακούσαμε ως παρατηρήσεις απόψε που το Συμβούλιο πραγματικά μπορεί να δεσμευτεί και δημόσια να πει ότι συμφωνεί με αυτέ τι παρατηρήσει. Είναι δέσμευση του Συμβουλίου, είναι δέσμευση που εκφράστηκε και με μια επιστολή που ε, απεστάλλει και όσον αφορά και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Και πρέπει λοιπόν στη διαπραγμάτευση που θα γίνει αυτό θα ληφθεί σίγουρα υπόψη. Συζητούμε λοιπόν μια διάμεση προσωρινή συμφωνία, προσωρινού χαρακτήρα, που βελτιώνει την μέχρι σήμερα κατάσταση. Συζητάμε για μια συμφωνία που έχει διάρκεια 9 μηνών. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβουλή και το Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε μια νέα συμφωνία. Τελική και τελεσίδικη καθοριστική συμφωνία. ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη όλα τα νόμιμα αιτήματα τα οποία διατύπωσε το Κοινοβούλιο απόψε. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε, το Συμβούλιο δεν μπορεί να αρνηθεί καθόλου τη συζήτηση που διεξήχθη εδώ. Δεν μπορούμε να αμελήσουμε ή να αγνοήσουμε ότι ήταν πολλέ οι επικριτικέ παρατηρήσει. Μεγάλη κριτική ασκήθηκε. Σίγουρα υπήρξαν κάποιε πιο καλά τεκμηριωμένες θέσει από άλλε τι επικρίσεις. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να ανοίξουμε μια περίοδο προβληματισμού, να τα ξαναδούμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεσμεύομαι και ζητώ χρόνο από πλευρά τη Ευρωβουλή. Ζητώ χρόνο χρόνο, είναι αυτονόητο αυτό βέβαια, για να υπάρξει διαβούλευση, να μπορέσω να σχολιάσω αυτά τα πράγματα με τους συναδέλφους του Συμβουλίου. Χρόνο για να τα σχολιάσω και να τα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρόνο επιπλέον ώστε να διαρευνήσουμε με τις ΗΠΑ τις δυνατότητες που νομίζω είναι πραγματικές και χειροπιαστές για να υπάρξει μια καλύτερη συμφωνία στο μέλλον. Χρόνο λοιπόν εν τέλει κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσω να ξανάρθω εδώ μπροστά σε αυτό το κοινοβούλιο σε κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες και να μπορέσω να επικυρώσω ενώπιόν σα ότι έχουμε τι βάσει στη διάθεσή μα για να υπάρξει μια τελική συμφωνία όπου τα μελήματα τα οποία εκφράσατε θα καλύπτονται επαρκώ. Είναι μια περίπτωση στι οποίε πάρα πολλέ φορέ συμπίπτει η τοποθέτησή σα με την τοποθέτηση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάλστρομ. Μπορεί να μην δουλεύει το μικρόφωνο. Όχι, δουλεύει, δουλεύει. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι η συζήτηση ήταν πολύ σημαντική και ακριβής διότι, και αυτό είναι σωστό διότι μιλούμε για σημαντικά θέματα την ασφάλεια των πολιτών αλλά ταυτόχρονα και ένα σύστημα που να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα. Το όπως είπε και το Συμβούλιο μπορεί να υπήρξαν και μερικές παρεξηγήσεις, μερικές όμως διαλύθηκαν, εξηγήθηκαν πρέπει να ξέρουμε όλοι γιατί έχουμε αυτή την ενδιάμεση προσωρινή συμφωνία. Για ποιο λόγο, για οποία αιτίαν. Διότι βρεθήκαμε μπροστά σε μια κατάσταση έλλειψης νομοθεσίας για τη μεταφορά των δεδομένων και γι' αυτό χρειάστηκε το Συμβούλιο και η Κομισιόν να αντιδράσουν σύντομα. εμπνεόμενοι από ορισμένου υπάρχοντες μηχανισμούς προστασίας δεδομένων και από τις ΗΠΑ. Ζητήσαμε παράλληλα να αποφεύγονται οι μεμονωμένες διμερείς συμφωνίες αλλά να γίνει μια πιο σφαιρική διευθέτηση. Είναι προσωρινή, ενδιάμεση αυτή η συμφωνία θα βελτιωθεί, έτσι προβλέπεται. Και το Συμβούλιο και η Κομισιόν σκοπεύουν να παίξει το ρόλο του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. χρειάζεται περισσότερη αποσαφήνιση για την αποθήκευση και την, των στοιχείων και το, τη, χρονική στιγμή κατά την οποία θα σβήνονται. Ο κύριος Λαμπρινίδης ρώτησε γιατί η Κομισιόν έπραξε τα πράγματα όπως τα έκανε. Μα εμείς είμαστε στα πράγματα εδώ και μερικές μέρες μόνον πρέπει πρώτα να βρούμε το χρόνο να το συζητήσουμε και μεταξύ μας πριν δοθεί πλήρης η διαπραγματευτική εντολή και θα το συζητήσουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού τόσο πρόσφατα διοριστήκαμε δεν μπορούτε να μας ζητάτε τέτοια πράγματα περισσότερα δηλαδή θα, ο κύριος Μπαρόσο σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Μπούσεκ θα δηλώνει ρητά ότι θα τα υποβάλουμε όλα αυτά εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τα γνωρίζετε όλα ε, Ίσως να είναι καλή ιδέα να μην γίνει αύριο η ψηφοφορία αλλά να αναβληθεί για να υπάρξει ο χρόνος να εξετάσετε όπως θέλετε και τη διαπραγματευτική εντολή και όλα τα σχετικά έγγραφα. Εμείς θέλουμε συνεργασία και με εσά και με το Συμβούλιο για να υπάρξει μια τελική, δεύτερη και πολύ πληρέστερη συμφωνία. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Συναδελφοί το η γαλάζια κάρτα δεν ισχύει κατά τη διάρκεια τη εισήγηση τη Επιτροπή και του Συμβουλίου. Αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Πρέπει να λάβουμε την αύριο απόφαση. Αν μπορώ λοιπόν, θέλω να σα ζητήσω να γίνει ίσως κατά παράβαση με το κανόνα ο κύριο Σούλφ και ο κύριο Λαμπρινίδης. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, πολύ σύντομοι να είστε. Τίποτα άλλο, γιατί θα μείνουμε εδώ άλλε δύο ώρε να συζητάμε το ίδιο θέμα. Ο κύριο Σούλτ, ναι κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σα άκουσα πολύ προσεκτικά. Όπω όλοι οι συνάδελφοι εξάλλου στην Ολομέλεια. Εσεί χρησιμοποίησατε τη διατύπωση και είπατε δώστε μας περισσότερο χρόνο ώστε να συζητήσω με τους συναδέλφους μου στο Συμβούλιο δώστε μου περισσότερο χρόνο ώστε να μπορέσω να επανέλθω με μια βελτιωμένη πρόταση συμφωνία. Σα ερωτώ λοιπόν πολύ χειροπιαστά και εξειδικευμένα. Αυτό που είπατε μπορώ να το εμεινεύσω έτσι ώστε ότι το Συμβούλιο δεν εμένει και δεν επιμένει σε αυτή τη συμφωνία πια και δεν επιμένει στην ψηφοφορία και στο αποτέλεσμα ώστε να έχετε χρόνο με τη ΣΥΠΑ να καταλήξετε σε μια καλύτερη διαπραγμάτευση για μια νέα καλύτερη συμφωνία. Κατάλαβα σωστά και ερμηνεύω σωστά ότι αυτό είπατε στην παρέμβασή σας. Ευχαριστώ. Κύριος Λαμπρινίδης, δεύτερη ερώτηση. Πολύ σύντομα και εσείς παρακαλώ. Okay. Το Συμβούλιο γνωρίζει το γεγονό ότι το SWIFT τα περασμένα χρόνια ούτε μία φορά δεν διαβίβασε συγκεκριμένα στοιχεία γιατί δεν μπορεί να τα ανασύρει και πάντοτε διαβιβάζει ε, χίδιν στοιχεία. Και ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις ΕΠΑ και το SWIFT ώστε αυτοί να εδράζουν στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε το σύνολο των στοιχείων που παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών να ελέγχονται μέσα εκεί. Επίσης δεν κάνει ούτε μία μικρή ε, υποχώρηση προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και οι Κομισιόν και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εξετάσουν πολύ σοβαρά το θέμα των χίδιν στοιχείων στην εντολή τη διαπραγματευτική. Ευχαριστώ. Δώσουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα για να μπορέσει να απαντήσει ο Προεδρεύων. Είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, λέει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θέλει για άλλη μια φορά να επιμείνει στη σημασία να μην διακοπεί η ροή χρηματοοικονομικών δεδομένων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΕΠΑ και αντίστροφα. Αλλά επίσης έχει συνειδητοποιήσει το Συμβούλιο ότι οι επιφυλάξεις, οι επικρίσεις, οι προτάσεις των κυρίων Ευρωβουλευτών πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού και εξέτασης. Και για αυτούς τους λόγους ζήτησα να μου δώσετε χρόνο για να προβληματιστούμε με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα διάφορα κράτη-μέλη στο σύνολό τους για την ανάγκη να ενταχθούν τέτοιου είδους στοιχεία στη νέα συμφωνία και αυτού του είδους ο προβληματισμός. Και ζήτησα περισσότερο χρόνο που νομίζω είναι πιο σημαντικό για να εξερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, αποκοινούμε τα κράτη-μέλη για τη βούληση που νομίζω ότι έχουν οι να ενταχθούν στη νέα τελική συμφωνία μεγάλος αριθμός από τα μέτρα αυτά για την πρόληψη, για τους όρους και προϋποθέσεις ε, και τα όρια που εξέφρασε το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να διέπουν αυτή τη συμφωνία. Εν τέλει, να αναζητηθεί καλύτερη ισορροπία στην τελική συμφωνία μεταξύ της ασφάλειας και της ελευθερίας ή των ελευθεριών που είναι τα θέματα που συζητάμε εδώ. Χρειαζόμαστε αυτό το χρόνο για να διερευνήσω αυτές τις δυνατότητες και να μπορέσω να προσέλθω στο Κοινοβούλιο σε μια τέτοια ολομέλεια προτού υπάρξει ε, η ε, ψηφοφορία. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η δέσμευση να μπορέσω να σας πω ότι έχουμε αυτή τη δέσμευση από τη ΣΥΠΑ. Υπάρχει η δέσμευση και σε σχέση με το Συμβούλιο να ενταχθούν αυτές οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νέα συμφωνία. Υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις η συζήτηση που θα είχαμε θα είναι διαφορετική από αυτή τη συζήτηση που έχουμε σήμερα απόψε εδώ. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Για να διατηρηθεί, ναι, η πολιτική ισορροπία σας καταλαβαίνω συνάδελφοι. Ο κύριος Βέμπερ και ο κύριος Πενέρα. Σύντομα όμως, πολύ σύντομα. Ναι, είναι μια μη συνηθισμένη συζήτηση. Από τα δεξιά λοιπόν δύο ερωτήσεις. Συνάδελφε, εγώ είμαι υπεύθυνο. Μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε αν θέλετε. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμο, Πρόεδρε, και ευχαριστώ που δίνετε την δυνατότητα να γίνει αυτό. Αν κατανοώ λοιπόν τα πράγματα σωστά, επειδή είναι πολύ ευαίσθητα θέματα αυτά τα οποία έτσι έντονα συζητούμε, τότε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου δεν μπορεί να μας διασφαλίσει ότι η ενισχύ αυτή η συμφωνία ε, αν αναβάλουμε θα, ε, δεν θα ισχύσει. Θα ισχύει λοιπόν. Και γι' αυτό θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Μπορεί να μας διασφαλίσει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου ότι για παράδειγμα μέσα σε ένα μήνα μια μακροπρόθεσμη διάρκεια συμφωνία θα είναι διαθέσιμη όπου οι ψηλότερες προδιαγραφές θα έχουν καθοριστεί ή λέει το Συμβούλιο παρόλα αυτά πρέπει να αναμείνουμε την εννεάμινη αυτή περίοδο μέχρι ότου εκπνεύσει αυτή η λεει το συμβουλιο παρολα αυτα πρεπει να αναμεινουμε την μηνη αυτη περιοδο μεχρι οτου εκπνευσει αυτη η περιοδο Τώρα, το θέμα τη αναβολή είναι κάτι πολύ δύσκολο για την Ευρωβουλή. Πρέπει να υπάρχουν σαφεί όροι και προποθέσει. Τι διασφαλίζει το Συμβούλιο για μια τέτοια πιθανή αναβολή, ώστε να γνωρίζουμε αύριο το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης που τον κανονισμό του σώματος ε, με γενναιόδωρο πνεύμα τον εφαρμόζεται και δίνεται τη δυνατότητα να παρέμουν δύο εκπρόσωποι από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και δύο από το ΕΛΚ. Η δική μου ερώτηση είναι η εξής, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Εσείς ε, θέσατε τον δάκτυλο στον τύπο των ύλων. Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης ε, και των συζητήσεων που έγιναν στο σώμα χρησιμοποιήθηκαν αξιοσέβαστα επιχειρήματα. Σέβομαι όλες τις παρεμβάσεις, αλλά οι λέξεις, τα λόγια όταν ε, εκφράζονται πρέπει να έχουν και μία πληροφορική ε, πληροφορία που μεταδίδουν και σίγουρα με εξέπληξε να βλέπω κάποιες τοποθετήσεις που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, το ατεκμηρίωτο δίνεται η εντύπωση ότι κανείς δεν διάβασε αυτή τη συμφωνία. Ότι πολύ λίγοι διάβασαν τη συμφωνία στην οποία ασκούν επικρίσεις. Γιατί αν την είχαν διαβάσει δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν με τέτοια επιχειρήματα όπως αυτά τα οποία ακούστηκαν. Έτσι λοιπόν πρόεδρε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι <clears throat> σε σχέση με αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος Μάνφρεντ Βέμπερ τι μπορεί να γίνει και σε σχέση με την κυρία την Πλάσερτ λέει σε σχέση με την επιστολή θα υπήρχαν όροι και ε, προϋποθέσεις ε, Ξέρετε ότι σε σχέση με την προσωρινή συμφωνία θα πρέπει να μπορεί να υπάρξει ε, παράλληλα η δυνατότητα διαπραγμάτευσης μιας νέας συμφωνίας. Όμως η κυρία η λέει και αυτό το οποίο ερωτά ο κύριος Μάφρετ Βέμπερ μπορεί να διασφαλίσει το Συμβούλιο σε σχέση με το Κοινοβούλιο τον Ιούνιο στην Επιτροπή και τον Ιούλιο στην Ολομέλεια να παρουσιαστεί το τελικό κείμενο με συμμετοχή της Ευρωβουλής στη νέα αυτή συμφωνία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μου ζητήσατε μια συγκεκριμένη εξειδίκευση χρονική και μία επί της ουσίας τοποθέτηση πιο χειροπιαστή. Σε σχέση με το χρόνο δεν είναι προφανές το ίδιο το να φέρει κανείς ε, στο σώμα τους όρους και προϋποθέσεις μιας τελικής ε, συμφωνίας που θα ισχύει ή με άλλο τρόπο να το πω, να προσκομίσω στο σώμα δέσμευση από πλευράς των ΗΠΑ για να ενταθούν κάποιες από τις παρεμβάσεις για τα μέτρα πρόληψης και τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Δεν είναι το ίδιο αυτό με το να υπάρξει μια νέα συμφωνία. Αν με ρωτάτε σε ένα μήνα αν θα είμαστε σε θέση να φέρω μια νέα συμφωνία στο σώμα, η απάντηση είναι όχι. Δεν είμαι σε θέση να το κάνω. Αν μου πείτε σε κάποιους λίγους μήνες μπορούμε να προσκομίσουμε στο σώμα το αποτέλεσμα κάποιων διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ με συμμετοχή πλέον της Ευρωβουλευτών Νομίζω ότι αυτό είναι πιο ουσιώδες και το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί αν πραγματικά όπως πιστεύει το Συμβούλιο θα έχουμε λόγους για να πούμε ότι η τελική συμφωνία θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή τη στιγμή, τότε η απάντησή μου είναι ναι. Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση υπό αυτούς όρους να το πετύχουμε. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο σας ζήτησα. Γι' αυτό δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρόταση της εισηγήτριας, που αληθεύει ότι είναι μια πρόταση που έχοντας δει τη γενική ατμόσφαιρα που επικρατούσε και τις πολλές παρεμβάσεις που υπήρχαν κατά της ε, προσυπογραφής της προσωρινής συμφωνίας, νομίζω τα πράγματα έχουν ως έχουν. Και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ρεαλιστικό, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, να ζητήσω χρόνο από την Ευρωβουλή, ώστε μέσα σε μια προθεσμία τριών μηνών να προσκομίσω εδώ προς συζήτηση στην Ευρωβουλή τα θεμέλια μιας συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ ή καλύτερα τα στοιχεία τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΠΑ, ΕΕ, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι πρέπει να ενταχθούν στην τελική συμφωνία που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση στη συνέχεια. Υπό αυτού του όρου ε, η συζήτηση θα ήταν τελείω διαφορετική, πιστεύω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Προεδρεύοντα. Την τελευταία λέξη στη συζήτηση την έχει η κυρία η η Ζανίν Χένι Πλάσκαρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Μπουζουτήλ και τον Προεδρεύοντα ιδιαίτερα ότι αν δεν χορηγήσουμε την έγκρισή μας αυτό δεν γίνεται γιατί δεν δεχόμαστε συμβιβασμό. Αυτό είναι τελείως λανθασμένο επιχείρημα. Υπάρχουν και άλλα νομικά εργαλεία και για την ε, έγκριση των μεταφορών δεδομένων δεν χρειάζεται να, περάσουμε, να περάσουν από εμά, αλλά το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε περισσότερο τους πολίτες. Θα έπρεπε να προσθέσω ότι η ενδιάμεση αυτή συμφωνία είναι εκβιαστική. Με συγχωρείτε που εκφράζομαι οργισμένα, αλλά νομίζω ότι το TFTP δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβαδίζει με, τα, με την ευρωπαϊκή παράδοση για τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Το έχω ξαναπεί και θέλω να το ακούσουν ξανά όλοι. Κανείς δεν αμφισβητεί τη την αναγκαιότητα να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ένωσης και ΕΠΑ ΕΕ ιδιαίτερα και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλά πρέπει να έχουμε δικούς μας στόχους. Και επομένως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαφωνούν από αυτού, ακόμη τουλάχιστον. Τέλος, το θέμα είναι θέμα ευθύνης της Ευρώπης και πρέπει να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση. Άκουσα προσεκτικά όσα είπατε και ότι ζητήσατε περισσότερο χρόνο. Και αυτό θα το ζητήσω από τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Μπορώ να το ζητήσω. Αλλά τα επιχειρήματά σας ήταν πολύ αδύνατα. Θα τη μεταφέρω. Θα το μεταφέρω το αίτημα αυτό αργότερα σήμερα στη διάσκεψη των Πρόεδρων για αναβολή της ψηφοφορίας. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι για τη συζήτηση, ήταν πολύ σημαντική. Δεν ξεπεράσαμε το χρόνο μας κατά περίπου 40 λεπτά, αλλά ήταν απαραίτητο. Αύριο στις 12 θα γίνει η ψηφοφορία, σας κατευχαριστώ. Λίγη εδώ η συζήτηση.